συστήματο τη Ένωση. Επ' αυτών των σημείων, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, προ... να φροντίσει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στου κανόνε που ισχύουν τώρα και αυτό να γίνει κατεπηγόντω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Καπούτο. Ο κύριο Μαριά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε την Τραπεζική Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί έχει αναλάβει την εποπτεία των συστημικών τραπεζών. Και όμως ο κύριος Δράγκη, ο οποίος ήταν εδώ, αναχώρησε δεν έμεινε σε αυτή τη συζήτηση να ακούσει τις παρατηρήσεις του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου παρότι ο ίδιος είπε ότι τον ενδιαφέρει η διαβούλευση. πάντως για τα κόκκινα δάνεια είπε ότι επί του πρακτέου η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να κάνει τίποτε. και όμως ο ίδιος ως ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα πιέζει τις τράπεζες στην ελλάδα προκειμένου να ξεπουλήσουν τα κόκκινα δάνεια να τα ξεπουλήσουν στα κοράκια σε τιμή τέτοια η οποία βεβαίως είναι πάρα πολύ φτηνή και εν συνεχεία τα κοράκια να αρπάξουν τα σπίτια των ελλήνων ενώ υπάρχει λύση στο θέμα αυτό. υπάρχει λύση την οποία έχουμε προτείνει η δημιουργία ενός ταμείου σωτηρίας δανειοληπτών προκειμένου να μην χάσουν οι έλληνες τα σπίτια τους. δυστυχώς δεν παρέμεινε εδώ ο κύριος δράγκη να ακούσει τους προβληματισμούς μας και να μπορέσει να έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. έχει πάρει τις αποφάσεις του και στα θέματα των κόκκινων δανείων. ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαριά. Κλείνει την διαδικασία αυτή και ο Σαφοζέρ. Ε, ε, θα ήθελα να μιλήσω για την ανευθυνότητά σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι, είστε ανεύθυνοι, γιατί τη στιγμή που οι τράπεζες δεν δανείζουν πια μεταξύ τους, και οι αγορές δεν έχουν πια εμπιστοσύνη στι Τράπεζε. εσείς θέλετε παρόλα αυτά να θεσπίσετε την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Είστε ανεύθυνοι λοιπόν γιατί δεν αναγνωρίζετε ότι η Νομισματική Ένωση δημιουργεί αυτή την τον ανεύθυνο δανεισμό γιατί πάντα κάποιο άλλο την πληρώνει. Και είστε ανεύθυνοι γιατί στην τελική ανάλυση θα πληρώσετε σπασμένα ο φορολογούμενος από το bailout περνάμε στο bail-in, ώστε οι ίδιοι οι φορολογούμενοι, οι ίδιοι οι πολίτες μέσω της συμμετοχή τους ή των καταθέσεων τους θα πληρώνουν. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσετε αυτή την ανευθυνότητα και οι τράπεζες, τα κράτη θα πρέπει να παρεθνικοποιήσουν τις κεντρικές τους τράπεζες, να αναλάβουν και πάλι την ευθύνη και να αποφύγουμε μελλοντικέ κρίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έκλεισε η διαδικασία προσέλκυσης προσοχή του Προέδρου Κάτσδιάη. Αλλά για να ολοκληρωθεί η συζήτηση θα δώσω το λόγο για μια ακόμη φορά, καταρχά στον Επίτροπο τον uh, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ εκ νέου κύριε Τόρβαλτς, έξοχη η έκθεσή σας. Άκουσα προσεκτικά στις παρεμβάσεις των, μελών. Αυτή η συζήτηση καταδεικνύει ότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι έχει σημασία η Τραπεζική Ένωση και έχει σημασία να υπάρχει ρυθμιστικό και υποπτικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στι τράπεζε να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, ασφαλίζοντα ότι το χρηματοστικό σύστημα είναι σταθερό και υγιέ. Yes, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να σημειώνουμε πρόοδο επί των χαρτοφυλακίων που έχουμε όσον αφορά τι χρηματοστικέ υπηρεσίε. Επίση, αυτή την τελευταία περίοδο πριν από τι εκλογέ, και βασιζόμαστε σε εσά να βοηθήσετε να εξασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε απτή πρόοδο για την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση, την Ένωση των Κεφαλαγορών και τελικά να έχουμε ισχυρή τραπεζική και νομισματική ένωση που θα είναι αρκετά ανθεκτική και να μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μελλοντική κρίση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επιτρόπε. Τη συζήτηση θα τον ολοκληρώσει εισηγητή, ο κύριο Τόρβαλ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή έχει αναδείξει τα βασικά στοιχεία της συζήτησης. Ναι, χρειαζόμαστε ένα σύστημα, ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων και επίσης θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να ξεπεράσουμε τον πόλεμο χαρακομμάτων που κάνουν μερικά κόμματα, πολιτικά κόμματα. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημά μας. Κύριε Βιέγκας, ανησυχείτε για τη μόχλευση. Μην ξεχνάτε όμως ότι τα ποσοστά μόχλευσης έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους και ηγητές. Θερμά ευχαριστώ για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Ήταν μεγάλη χαρά που διοργανώσαμε αυτή τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ελπίζω, χάρη σε αυτή τη συζήτηση, να φανεί η ακολουθητέα πορεία και να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο γιατί υποσχέθηκε ότι θα υποβάλει ως ονόπο τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Τόρβαλ. Σε η συζήτηση αύριο θα ψηφίσουμε. Και περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησιά διάταξη ε, Έκθεση των συναδέλφων ε, Φερνάντεθ και Γουαρτάντες και Γουαλτιέρη, Θέσπιση του προγράμματο InvestEU. Οι εισηγητέ θα πάρουν πρώτα το λόγο. Τέσσερα λεπτά ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και να τους πω ότι στην κατάλληλη στιγμή σημειώνουμε πρόοδο για αυτό το InvestEU, το πρόγραμμα που συνενώνει 13 χρηματοδοτικά μέσα. Θα εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη απλούστευση και θα, θα πληρώσει κάποια κενά της αγοράς. Και έχει τέσσερις άξονες, τις υποδομές, την έρευνα και την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τον κοινωνικό πυλώνα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια συνέχεια και συμπληρωματικότητα των προηγούμενων χρηματοδοτικών μέσων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του επενδυτικού σχεδίου Juncker. Και με το πρόγραμμα αυτό ε, υλοποιήσαμε 1,2 εκατομμύρια ε, ε, Θέσει απασχόληση και υποστηρίξαμε 200.000 ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βοηθά την οικονομική ανάπτυξη, στηρίζει τι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τι φιλοδοξίε του επενδυτικού σχεδίου τι συνεχίζει και τι αναβαθμίζει το πρόγραμμα InvestEU. Και για αυτά τα τρία χρηματοδοτικά μέσα που συνενώνει το InvestEU προτείνουμε ενίσχυση των εγγύησεων ώστε να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας. Έχουμε μία μικρή διαφορά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επ' ευκαιρία θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ και να χαιρετήσω τον Αντιπρόεδρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 650 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς προτείνουμε 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, θεωρούμε, όπως είναι προφανές, ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι απόλυτα εξασφαλισμένες και οι στόχοι για το περιβάλλον, για το κλίμα, για την στρατηγική ε, που θέλουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει όλα αυτά να διασφαλιστούν και να αποφύγουμε φυσικά και τους αποκλεισμούς. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρειάζεται μια ασφάλεια δικαίου, ώστε να δίνει το 75% της εγγύησης και οι άλλες τράπεζες ε, πρόθεσης, εθνικές ε, και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να έχουν πρόσβαση στο υπόλοιπο 25%. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό, το InvestEU, να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, στην εδαφική συνοχή, αλλά και στην οικονομική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό η γεωγραφική ισορροπία είναι κάτι πολύ σημαντικό για το InvestEU. Επίσης, έχουμε τη σημαντική πλατφόρμα ε, για την παροχή συμβουλών, επενδυτικών συμβουλών. Αυτή η πλατφόρμα θα ενισχυθεί ώστε και τα περιφερειακά προγράμματα και τα σχέδια των πιο απομακρυσμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πρόσβαση στο InvestEU και στη χρηματοδότησή του. Και να φροντίσουμε και τα πιο μικρής εμβέλειας σχέδια. Θα πρέπει να υπάρχουν πλατφόρμες επενδυτικές και αυτή ε, η πλατφόρμα παροχής συμβουλών, αυτό το δίκτυο παροχής συμβουλών, καλό θα ήταν να έχει μια δυναμική προσέγγιση και προορατική. Στην πρότασή μας ε, προτείνουμε κάποια απλούστευση και τη διακυβέρνηση. Επίσης, ό,τι αφορά την προσθετικότητα, θέλουμε να διατηρηθεί και βέβαια να την προσαρμόσουμε στη νέα πραγματικότητα και ε, στη συγχώνευση αυτών των 13 χρηματοδοτικών μέσων δεν θα πρέπει επίση να ξεχνούμε τις κοινωνικέ επενδύσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους και ηγητές, τον συνεισηγητή μου φυσικά, τον κύριο Γουαλτιέρη. που είναι από τους σοσιαλιστές, να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ότμαρ Κάρα για την πολύ χρήσιμη συνεισφορά του και να ευχαριστήσω και του λοιπούς και που συμμετείχαν στη διαμόρφωση της έκθεσης για το πρόγραμμα InvestEU που θα συμβάλλει τα μάλα στην οικονομική ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φερνάντες. Τώρα ο συνεισηγητής ε, κύριος Γκουαλτιέρη επίσης για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φερνάντες και όλους τους κοιόδης εισηγητές. Ήταν έξοχη η συνεργασία μας. Η κρίση του 2008 προξένησε άνευ προηγουμένου πτώση των επενδύσεων και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια οι συνθήκε για τι επενδύσει στην Ευρώπη βελτιώθηκαν χάρη σε μια οικονομική κατάσταση που είναι πιο ευνοϊκή, χάρη στην ευελιξία όσον αφορά την ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητα, χάρη σε νέε πρωτοβουλίε όπω αυτή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τι Επενδύσει, στρατηγικέ επενδύσει, αλλά όγκο των επενδύσεων στην Ευρώπη παραμένει κάτω από τον μέσο όρο που είχαμε πετύχει στη δεκαετία πριν από την κρίση. Τα νέα και πιο μεγάλα κενά έχουν ανοίξει στους τομείς που συνδέονται με την καινοτομία, με τις φυσικές και κοινωνικές υποδομές και την αλλαγή του κλίματος. Αυτή η κατάσταση μας ανησυχεί όσον αφορά το μέλλον της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής της Ευρώπης για την ανάπτυξη της μακροπρόθεσμα και για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό είναι θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνοντα τη θέσπιση ενό προγράμματο Invest EU ήθελε όχι μόνο να ανανεώσει αλλά και να αντικοπήσει την υποστήριξη των επενδύσεων. Το Invest EU δεν είναι μόνο ένα εργαλείο που, που συνεχίζει την θετική εμπειρία του FACE και άλλων ε, προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν αυτά τα χρόνια. Πέρα από την ενίσχυση, την περαιτέρω ενίσχυση, την υποστήριξη των μισομεσαίων επιχειρήσεων, ε, τι βιώσιμε υποδομέ, την έρευνα και την ανάπτυξη, αυτό το πρόγραμμα θέλει να αντιμετωπίσει τα τεράστια κενά που υπάρχουν στι υποδομέ κοινωνικέ που αναφέρθηκε στην έκθεση ε, το, του, τον Ιανουάριο Task Force που εξετάζει το θέμα αυτό και για το ότι θα στο τομέα της παιδείας, της υγείας και των κοινωνικών κτηρίων θα πραγματοποιούνται τα προγράμματα. Πρωταρχικός στόχος του InvestEU είναι να καλύπτει επενδυτικά κενά στους τομείς και τους γεωγραφικές περιοχές που υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Και για να το πετύχει αυτό παρενέβη με σειρά τροποποίησεων βελτιωτικών το Κοινοβούλιο σχετικά με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν πρώτης Είπαμε ότι το κόστος της εγγύσης για την πρόθεση των επενδύσεων θα πρέπει αποκλειστικά να συνδέεται με τα χαρακτηριστικά και τον κίνδυνο των επιχειρήσεων που αδρομολογούνται και ποιες θετικές συνθήκες θα μπορούν να εφαρμόζονται για να δημιουργούνται επενδυτικέ πλατφόρμε, για να διευκολύνονται οι επενδύσει στου τομεί όπου τα επενδυτικά κενά είναι μεγαλύτερα ή για να ανθαρρύνουμε παρεμβάσει στου τομεί εκείνου όπου υπάρχει ανάγκη επενδύσεων, ε, μεγαλύτερη ανάγκη επενδύσεων. Δεύτερον, πέρα από το επαναλαμβάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τάπεζα Επενδύσεων θα είναι οικονομικό εταίρο, οικονομικό βασικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό του InvestEU, Αξιολογήσαμε και το σημαντικό ρόλο που έχουν οι τράπεζε, οι εθνικέ προθήσεων και χρηματοδοτήσεω έργων επενδυτικών. Ε, οι εθνικέ αυτέ επενδυτικέ τράπεζε μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση ε, στι ευρωπαϊκέ εγγύσει. Αυτό θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερε δυνατότητε χρηματοδοτήσεω διαφόρων έργων ε, που θα έχουν θετικές επιπτώσεις αφορά τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, αποφασίσαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν μόνο τη δυνατότητα να δίνουν ένα μέρος των πόρων που δίνουν για την πολιτική συνοχή για αυτό το σκοπό, αλλά θα μπορούν να συμβάλλουν και με πρόσθετους πόρους που καταρχήν θα θεωρούνται σαν one-off, σαν εφάπαξ συνδρομή όσον αφορά την κάλυψη των διαθροτικών έλλειμμάτων που συμπεριλαμβάνονται σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Είναι ισορροπημένη η έκθεση και, και όπως και το τμήμα που λέει ότι τουλάχιστον 65% των επενδύσεων στα πλαίσια των βιωσίμων υποδομών θα συμβάλλουν να πετύχουμε τους ε, καθοριστέντες στόχους των συμφωνίας των Παρισίων για το περιβάλλον και το κλίμα. Ζητώ να παραμείνει το κείμενο ψηφίστηκε από την Επιτροπή Οίκων στο τομέα αυτό όσον αφορά το όριο του 65%. Με αυτό το κείμενο πιστεύω ότι δίνουμε μια συγκεκριμένη απάντηση σε εκείνους που θέλουν η Ευρώπη να κάνει περισσότερα για τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και την εργασία. Ευχαριστώ και τον κύριο Γκουαλτιέρη. Ο κύριος Κέλλη έχει τώρα το λόγο. Ένα λεπτό. Ε, το InvestEU είναι εμβληματικό πρόγραμμα ε, στο πλαίσιο του νέου προπολογισμού για το 2021-2027. 650 δι θα διατεθούν για επενδύσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έτσι ε, είναι ένα παράδειγμα που μα δείχνει πόσο αποτελεσματικέ είναι επενδύσεις, μεγαλύτερε επενδύσει, με λιγότερο κόστο για του φορολογουμένου. Τα τελευταία δύο χρόνια παρακολούθησα πολλά τέτοια επενδυτικά προγράμματα που οργανώθηκαν στην περιφέρειά μου από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Κατάιν ήταν εκεί, μεταξύ άλλων. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό για το InvestEU ε, και γνωρίζω ότι τουλάχιστον στη δική μου περιφέρεια είναι κάτι που το περιμένουν ε, με τεράστια όρεξη οι εργοδότες και επιχειρηματίες και ελπίζουμε να τονώσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή Ήτρε είναι κάτι που το περιλάβαμε στην γνωμοδότησή μας και το δέχτηκαν όλε τις πολιτικές ομάδες και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα. Δεν μιλάμε μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ανεξάρτητο τρόπο ε, να συγκεντρώνουν κεφάλαιο. Μιλάμε κυρίως για τις μικρές. Αυτές πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο και χαίρομαι που τελικά το κάνουμε. Ολοκληρώνοντας, ήθελα να πω πώς θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε και στο συνολικότερο πλαίσιο του τι γίνεται σήμερα στο Westminster. Νομίζω ότι δεν έχω ολοκληρώσει. Δεν είχα 1,5 λεπτό. Α, ένα λεπτό είχα. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι αυτό είναι το απόλυτο αντίδοτο στο Brexit, γιατί θα βοηθήσει τι επιχείρησει που θα πληγούν να, να έχουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση ώστε να επιβιώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλ. Είχατε δυστυχώς ένα λεπτό στην ε, διάθεσή σας. Ε, συνήθως ε, πέφτεται μέσα αυτή τη φορά, όμω δεν είχατε παραπάνω. Δεν μπορώ να επιτρέψω τι μπλε Επόμενο Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, κύριος Βαντενκάμπ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο συνεισηγητές και τους και για γιατί πολύ αξιόλογη τους πρόταση και για το ότι έφερα σε αίσιο πέρας ε, αυτή τη σημαντική συζήτηση. Αυτό χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα για τον τομέα των μεταφορών. Και ιδιαίτερα όταν μιλούμε για την ε, κατασκευή ε, αυτοκινητοδρόμων και οδικού δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση για τις υποδομές στις οδικές μεταφορές, μεταξύ άλλων. Επίσης, ας μην ξεχνάμε και τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Το επισήμαναν και η γνωμοδοτήση Επιτροπής ΕΚΟΝ και Περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε και ιδιωτικές επενδύσεις βέβαια, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι ό,τι αφορά του περιβαλλοντικού μα στόχου. Πρέπει να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μα εκεί. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Κατάινεν. Κύριε Πρόεδρε, είμαι βουλευτή, βουλευτέ, με μεγάλη χαρά συμμετέχω στη συζήτηση και με μεγάλη χαρά βλέπω και τόσου πολλού συναδέλφου παρόντε ε, ε, συναδέλφους οι οποίοι ε, θέλησαν να εφαρμόσουν το έτσι στις ε, περιφερειές τους, βλέποντας τι μπορεί να γίνει με τις επενδυτικές υπηρεσίε τη... και προσπάθησαν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση. Εξού και η επιτυχία του έτσι μέχρι τώρα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την πολύ καλή αυτή αρχική επιτυχημένη λύση με το έτσι. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την πρόταση για το InvestEU. Θέλω να ευχαριστήσω το σώμα που στην ε, θητεία αυτή υποστήριξη τις προτάσεις της Κομισιόν για τις επενδύσεις. Όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ε, στα τέλη του 2014 είχαν πέσει οι επενδύσεις κατά 15% λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και χρειάστηκε να ληφθούν ε, συνολικά μέτρα και δράσεις για να κλείσει το επενδυτικό κενό και για να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη και στην οικονομία της Ένωσης και στις δυνατότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να δώσουν αποτέλεσματα στους πολίτες. Το Invest EU ε, τώρα είναι η απάντηση στην κατάσταση. Πρώτα, βέβαια, είχαμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που ήταν το πρώτο βήμα. Έχουν ε, λοιπόν βελτιωθεί έκτοτε οι επενδύσεις. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει επενδυτικό κενό, ιδίως σε κοινωνικές υποδομές και υποδομές ε, στην περιβαλλοντική μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση. Επομένως για το προσεχές πολιετές μεσονομικό πλαίσιο έχουμε την ενιαία αυτή πολιτική για την υποστήριξη των επενδύσεων, ε, το Ταμείο EU, ε, InvestEU, που θα συμπεριλαμβάνει 13 κεντρικώς διαχειριζόμενα μέσα και το ΕΤΣΕ. 38 δις θα είναι ο προϋπολογισμός. Θα έχει έντονη εστίαση στις πολιτικές. Στρατηγικός εταίρος λοιπόν η Κομισιόν και ευπρόσδεκτη και άλλοι εταίροι όπως είναι η Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλοι εθνικοί και διεθνεί ε, τραπεζικοί φορεί. Χαιρετίζουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το InvestEU. Η έκθεση πραγματεύεται σημαντικά ζητήματα ε, αλλά σε ευρεία βάση συμφωνεί και με τι προτάσει τη Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τι προτινόμενε αλλαγέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή να εξετάσει τι αλλαγέ που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση και ιδίω αυτέ που κάνουν λόγο για αύξηση ε, τη αυτονομία τη ε, σχετική επενδυτική επιτροπή και διασφάλιση των πολιτικών τη Κομισιόν. Υπήρξαν κάποιε ανησυχίε για το ρόλο τη ΕΤΕΠ στο πλαίσιο του InvestEU σε σχέση με το ΕΤΣΑ. Θέλω να σα πω πω και η ε, Κομισιόν και η ΕΤΕΠ έχει, έχουν καταλήξει ε, σε συμφωνία για αυτό το 75%. Η εταιρική σχέση θα βοηθήσει να αξιοποιηθεί τα μάλα η εμπειρία της ε, ΕΤΕΠ για τις διάφορες συναλλαγές, για την παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών κινδύνων και για την εφαρμογή του ε, προγράμματος φυσικά οι συνομοθέτε θα έχουν τον έλεγχο. Κάποιε από τι τροπολογίε σα σχετίζονται με την ευρύτερη συζήτηση για το πολιετέ, όπω το συνολικό ποσό τη εγγύηση και το σύμφωνο για το κλίμα. Σημειώνουμε τις προτάσεις. Είναι μια μαρτυρία του πόσο δεσμευμένο, πόσο προσιλωμένο είναι το Κοινοβούλιο σε μια ισχυρή ένωση με ένα ισχυρό προπολογισμό και την εφαρμογή των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της COP21. Ε, Επίσης θέλουμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τις ε, πολύ μεγάλες προσπάθειες ε, του εισηγητού, των εισηγητών και όλων των άλλων συναδέλφων. Κατάφεραν να συμφωνήσουν μέσα σε ένα πολύ φιλόδοξο χρόνο διάγραμμα ώστε πριν τι ευρωεκλογέ να έχουμε καταλήξει. Ελπίζω αυτέ οι άκουνε προσπάθειε ε, να αντικατοπτριστούν και στην αυριανή ψηφοφορία. Τώρα πλέον το Συμβούλιο είναι αυτό που πρέπει να αναβαθμίσει τι προσπάθειέ του, ώστε να φτάσουμε σε μια γενική προσέγγιση που θα είναι αμερόληπτη, αντικειμενική, θα επιτρέψει την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Επιτροπέ Κατάινεν. Τώρα ο κύριο Μπέλετ, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Eh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ας συγκρίνουμε ε, το InvestEU με το τρέχον ε, Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Βλέπουμε ότι ε, οι επενδύσεις είναι περισσότερες για την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή ασφάλεια Ελπίζουμε να αυξηθεί το ποσοστό που τώρα είναι 15% και να δώσουμε έμφαση στη βιωσιμότητα και το περιβάλλον. Αυτό θα πρέπει να είναι το κοινό χαρακτηριστικό και ένα είδος μη του για όλα τα προγράμματα του InvestEU και όλα τα σχέδια που θα χρηματοδοτήσει. Επίσης, θα πρέπει να περιορίσουμε την παραγωγή άνθρακα με γνώμονα φυσικά τη βιωσιμότητα. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε καλά όλα αυτά τα εργαλεία και όπως είπε ο κύριος Κέλλη, το πρόγραμμα InvestEU είναι εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα σημαντικότερα προγράμματά μας για να έχουμε βιώσιμη ενέργεια και σε προσιτές τιμές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπέλετ. Κυρία Βέστφαλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, πιστεύω πως το InvestEU είναι ένα καλό πρόγραμμα και πράγματι θεωρώ ότι η έκθεση των ε, συνεισηγητών ε, βελτιώνει το πρόγραμμα. Αν μου επιτρέπετε όμως ε, να ρίξω λίγο νερό στο κρασί ως υπεύθυνη για την περιφερική πολιτική. Κατά την άποψή μου, τα διευθυντικά ταμεία με την αποκέντρωση, με την επιμερισμένη διαχείριση είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το InvestEU. Τα διευθυντικά ταμεία, επομένω, είναι αυτά τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή όλων των Ευρωπαίων πολιτών, διότι δίνουν θέσει εργασία στι περιφέρειε, βελτιώνουν τι υποδομέ, αντιμετωπίζουν την αλλαγή του κλίματο, στηρίζουν τι επιχειρήσει και τα πανεπιστήμια και θα πρέπει οι ενισχύσει αυτές να συνεχιστούν, ακόμη κι αν περικοπεί ο προπολογισμό. Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν συμφωνώ με την ιδέα τα διαρθρωτικά ταμεία να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του InvestEU, αλλά λέω ναι ε, στην ιδέα να έχουμε συνέργειες. Λέω όμως ε, όχι ε, στο να υπάρξει μια σύγχυση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση αυτών των δύο εργαλείων. Τζαμπάσκι τώρα για να... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αντιπροσωπεύω εδώ την Επιτροπή Πολιτισμού. Εμείς υπογραμμίσαμε την ανάγκη για συμπροματικές επενδύσεις για την νεολαία και για τον πολιτισμό. Οι τροπολογίες μας θα βοηθήσουν το να διαφυλάξουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά Ξέρετε ότι έχουμε μοναδική πολιτιστική κληρονομιά, μοναδική στον κόσμο. Πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές, διότι αλλάζει ραγδαία ο κόσμος και εμφανίζονται παντού νέες τεχνολογίες. Είμαι σίγουρος ότι το InvestEU θα προωθήσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πρέπει όμως να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε και την ταυτότητά μας πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι η εθνική ταυτότητα και ο εθνικό πολιτισμός, η εθνική κουλτούρα είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Κάθε περιοχή, κάθε χώρα θα πρέπει να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τους πόρους του Invest EU, έτσι θα μπορέσουμε να διασώσουμε και να διαφυλάξουμε την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσαμπάσκη. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο συνάδελφος Κάρας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι από την αρχή της ε, θητείας αυτής αγωνίστηκαν για ενισχύση των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδύσεις που σίγουρα πρέπει να κινητοποιηθούν και αυτό δεν είναι κούρσα ταχύτητας αλλά μαραθώνιος. Ε, και νομίζω βήμα το βήμα ε, μάθαμε πράγματα και βελτιωθήκαμε έγινε αυτή η επίθεση, αν θέλετε, η επενδυτική κατά την τη θητεία με το ΕΤΣΕ και με το ΕΤΣΙ νούμερο 2 μέχρι το 2020 ε, που επιμηκύνθηκε και βελτιώθηκε η κατάσταση. Συνέχισε και η επενδυτική, αν θέλετε, επίθεση σε τρίτες χώρες, κυρίως αφρικανικές ε, και με την νέα αυτή πρωτοβουλία, το Invest EU, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι την επόμενη επταετία να έχουμε 700, εκατομμύρια ευρώ ε, τα οποία θα βοηθήσουν ε, τις επενδύσεις, τη μείωση της ε, γραφειοκρατίας και θα ενισχύσουν, θα συγκεντρώσουν τις ενισχύσεις, θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δούμε ακριβώς ε, τι γίνεται και με την εγγύηση, ε, το μέσο αυτό και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σίγουρα η ε, διαφάνεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και εφαρμογή των στόχων για το κλίμα. Αυτό είναι ο συνολικός μας στόχος και έτσι πιστεύω θα έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για ανάπτυξη, για απασχόληση και περισσότερες επενδύσεις στην Παγκένωση. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίσουμε τη συζήτηση. Κυρία Γκαρθιαθάμπαλου Ρουμπιάλ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους συνεισηγητές Γουαλτιέρη και Φερνάντες ε, για το πολύ σημαντικό έργο που υλοποίησαν. Φυσικά ξεκινάμε από μια καλή αφετηρία, την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στην συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χάρη στους συνεισηγητές και τους κοιόδης συγητές των πολιτικών ομάδων, βελτιώσαμε την αρχική πρόταση. Από την αρχή της οικονομικής κρίσης, για τους σοσιαλιστές, προτεραιότητα ήταν ένα σχέδιο ε, επενδύσεων για να βελτιωθούν οι οικονομίες, αλλά με το σωστό τρόπο και μέσω μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Και μάλιστα ήδη ασχοληθήκαμε με το πρώτο επενδυτικό σχέδιο, το σχέδιο Juncker για τις ε, στρατηγικές επενδύσεις και ε, ασχοληθήκαμε και το δεύτερο επενδυτικό σχέδιο Juncker, τη διεύρυνση του ΕΦΣΥ και είχαμε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Με το InvestEU στηριζόμαστε όχι στα μέχρι τώρα θετικά αποτελέσματα και την εμπειρία του προηγούμενου σχεδίου στρατηγικών επενδύσεων, αλλά συνδυάζουμε και χρηματοδοτικά μέσα που ενέπτασε σε διαφορετικά προγράμματα. Επίση, με τη συγχώνευση αυτή θα έχουμε ένα πολύ πιο ελαστικό, αποτελεσματικό και απλό μέσο με καλύτερο αντίκτυπο. Επίση, θέλουμε περίπου 700 δισεκατομμύρια ευρώ κινητοποίηση χάρη στον Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό προπολογισμό προκειμένου να γίνουν επενδύσει, ώστε να επιτύχουμε μια ευφύ ανάπτυξη επενδύοντα στη γνώση, σε βιώσιμε υποδομέ ή στη βελτίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη βελτίωση τη πρόσβασή του στη δανειοδότηση. Επίση, θέλουμε να βελτιώσουμε και τι κοινωνικέ υποδομέ και να δώσουμε μια όθηση στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών να δώσουμε ιδιαίτερο ρόλο στι εθνικέ περιφερειακέ περιφερειακές ε, τράπεζες Θα δημιουργήσουν πολύ θετικέ συνέργειε ε, προκειμένου να προσαρμοστούν οι επενδύσει στις ιδιαίτερε ανάγκε των περιφερειών. Γι' αυτό α ξεκινήσουμε αμέσω τις διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Ελπίζω να καταλήξουμε σε θετική συμφωνία με βάση αυτά που θα ψηφίσουμε αύριο, ε, δηλαδή με βάση του στόχου μα, αλλά κυρίω με βάση τον προπολογισμό που θα ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλμελ έχει τώρα το λόγο. Για 1,5 λεπτό. Από την ομάδα ECR. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με το InvestEU στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ακόμα μια προσπάθεια με τις δαπάνες, τις νέες, να ε, λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης υποδομών. Ούτε θα πετύχει, ε, ούτε και έχει πετύχει κατά το παρελθόν αυτή η προσπάθεια. Το θέμα είναι να γίνουν αναλύσεις και να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα. Αν όμως λέμε ε, θέλουμε περισσότερες επενδύσεις, το κάνουμε σαν να είναι όλες οι επενδύσεις καλές. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Μόνο αν είναι βιώσιμα τα αποτελέσματά του είναι επενδύσει. Θα πρέπει λοιπόν επιτέλου να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αρθεί πάνω από τις ιδιωτικές επενδύσεις ή την ιδιωτική οικονομία συγκεκριμένα. Χρειαζόμαστε ιδιωτικές επενδύσεις και σίγουρα υπάρχει χρήμα. Χρήμα υπάρχει αλλά πρέπει να επενδυθεί. Άλλα προβλήματα έχουμε ε, και δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι να τροφοδοτήσουμε χρήματα την ιδιωτική οικονομία. Το ίδιο ισχύει με το σχέδιο το επενδυτικό του Juncker, το έτσι. Δηλαδή χρηματοδοτούμε κάποια project χωρίς να ξέρουμε τι αποτελέσματα θα έχουν και χωρίς να ε, μπορούμε να μετρήσουμε τελικά τα αποτελέσματα. Και έτσι θα έχουμε λάθος ε, ε, χρηματοδοτήσει. Δεν θα κάνουμε καλός πολίτες. Και αυτό το οποίο θα χρειαζόταν, αν θέλουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, θα ήταν μια μεταρρύθμιση του νομίζω νομίσματος, του ευρώ. Γιατί πραγματικά ε, ουσιαστικά κάνει πράγματα, μάλλον εξισώνει πράγματα που δεν πρέπει να εξισώνονται και ε, αυτό ε, θα βελτίωνε την οικονομία μας αν αλλάζαμε την κατάσταση πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρος. Και τώρα θα δώσω το λόγο για δύο λεπτά στον κύριο Τόρβαλ, συγγνώμη τη Άλντε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε και εσείς, κούσουναμ στη γλώσσα σας. Ευχαριστώ. Επίτροπε Κατάινεν, εδώ και χρόνια, όταν ξεκινήσαμε αυτό το μακρύ ταξίδι, ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας όσον αφορά το σχέδιο Juncker. Πολλοί από εμά ήμασταν αρκετά διστακτικοί τότε. Διρωτώμεθα κατά πόσο θα έδινε την κατάλληλη όθηση. Έχουμε μάθει πολλά, είμαστε σοφότεροι τώρα και βλέπουμε ότι οι τροχοί γυρίζουν. Βέβαια, υπάρχουν πολλά προβλήματα που μας περιμένουν, πολλές προκλήσεις, προσπαθώντας να κάνουμε το δεύτερο και το τρίτο βήμα. Το InvestEU είναι ένα άλλο είδος ποδηλάτου, ούτως υπήν, σε σχέση με το FC1 και το FC2. υπησέρχονται και εξωτερικές δυνάμεις που δεν καλύπτονται από τα θεσμικά όργανα, που δεν είναι στο πλαίσιο θεσμικών οργάνων. Όταν συζητούμε αυτά τα θέματα στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, φαίνεται σαν να υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το αν θα καταφέρουμε πραγματικά τους εξωτερικούς φορείς να τους εντάξουμε, να συμβάλλουν στην προσπάθεια. Πάντα ακολουθούμε μια εθνική προσέγγιση στα πράγματα. Και όταν έχουμε την εθνική οπτική γωνία, όταν συζητάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αν σκεφτόμαστε σαν ένα κράτος, αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο εγχείρημα αυτό, να ευχαριστήσουμε τους εισηγητές για τη δουλειά τους και κάνουμε ένα μεγάλο βήμα πρόοδου σήμερα και αύριο. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να μας ακολουθήσει μαζί με το Κοινοβούλιο να κινηθεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν γίνει αυτό θα, είμαστε πολύ, θα είναι όλα πολύ καλύτερα για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γκίγκολτ για 1,5 λεπτό εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι ήταν κατεπίγουσα η ανάγκη η Ένωση να κινηθεί πιο δραστηρία για να αυξήσει τις ε, επενδύσεις. Γι' αυτό ευπρόσδεκτη η προσπάθεια για το έύση το αρχικό. Είδαμε τα κενά που υπήρχαν. Μάθαμε από τις ελλείψεις. Και τώρα έχουμε μια νέα πρόταση. Η Ένωση πρέπει να είναι τολμηρότερη, να αυξήσει τις επενδύσεις. Και το πρόγραμμα Invest EU περί αυτού πρόκειται. Ταυτόχρονα να τονίσω ότι η καλή επένδυση είναι μόνο η βιώσιμη επένδυση. Μόνο η επένδυση που αντλεί τα μαθήματα από την κρίση του κλίματος είναι μια καλή επένδυση. Γι' αυτό ήταν θετικό το ότι ο συμβιβασμός που απορρέει από την καθήλια αρμόδια επιτροπή για την αύξηση του ποσοστού βιωσίμων επενδύσεων στο παράθυρο των επενδύσεων στο 65% είναι σημαντική. Είναι σημαντικό η ομάδα μας να διατηρήσει αυτή την πρόταση το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, πιστεύουμε ένθερμα ότι στατιωτικοί και πολιτικοί στόχοι στους προπολογισμού πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς. Και αυτή η αρχή θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και στην Ολομέλεια, στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια και βασίζομαι στους συνεισηγητέ να ακολουθήσουν τις αρχικές συμβαστικέ λύσεις και να μην αλλάξουν κατεύθυνση στην Ολομέλεια και έτσι να μην μπορούμε να πετύχουμε μια πανευρωπαϊκή ε, πλειοψηφία, κάτι το οποίο αξίζει αυτή η πρόταση κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κ. Παπαδημούλης έχει το λόγο. Όπως είπε και ο Επίτροπος Κατάινεν, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενίσχυση των επενδύσεων. Είμαστε ακόμη αρκετά πίσω από το επίπεδο των επενδύσεων προ-κρίσης. Επομένως, τα βήματα που γίνονται με το Investing You κατά την άποψη της πολιτικής μας ομάδας, δεν είναι αρκετά. Είναι γεγονός ότι η πρόταση που φέρνει το ευρωκοινοβούλιο βελτιώνει την αρχική πρόταση της κομισιόν σε αρκετά σημεία. εντοπίζω όμως κάποια αρνητικά και κάποιους κινδύνους. υπάρχει ο κίνδυνος το investeu να αφαιρέσει κονδύλια από το ταμείο συνοχής και αυτό θα είναι απαράδεκτο όταν έχουμε ήδη μείωση των κονδυλίων συνοχής στην πρόταση της κομισιόν για το νέο πολιετές πλαίσιο. και ο δεύτερος κίνδυνος είναι να αδικηθούν οι πραγματικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς θα επιμείνουμε περισσότερες επενδύσεις και ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη αποεπένδυση και σε αυτές τις περιοχές που έχουν υποφέρει περισσότερο από την ύφεση. Σας ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κόμπερν έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Uh, λοιπόν, τώρα το InvestEU επενδύει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα χειρίζεται σε κεντρικό επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να θυμηθούμε δύο πράγματα. Πρώτο, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρήματα προέρχονται από το φορολογούμενο και είναι χρήματα φορολογουμένων. Δεύτερον, θα πρέπει Επιχειρήσει που επενδύουν τα χρήματα του φορολογουμένων να θεωρηθεί ότι αυτά τα χρήματα είναι επιδότηση και στευλώνεται αγορά στην οποία βασίζονται οι φορολογούμενοι. Είτε είναι καταναλωτές, είτε είναι επενδυτές, είτε είναι και τα δύο. Οι κανόνες περικρατικών ενισχύσεων ήθελαν να εφαρμόσουν ισότιμους όρου όσον αφορά τη χρήση επιδοτήσεων. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θεσπίσει κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα ήταν ισότιμη όρια αν στη μεταβατική περίοδο ισχύουν αυτά. Διότι η διαδικασία έγκρισης προβλέπει ότι καλύπτει επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά όχι τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Ίσως θα πείτε ότι είμαστε στο τέλος της σειράς. Δεν θα έπρεπε να είναι κάτι μειονεκτικό. Ο Oliver Twist ήταν στο πίσω μέρος της ουράς για το επιθετούμενο φαγητό που έπαιρνε και το να ζητήσει περισσότερα δεν τον βοήθησε. Για να ξεφύγουμε τώρα, ε, ξεφύγαμε από το 19ο αιώνα και την κατάσταση αυτή και θα πρέπει να το κάνουν αυτό και οι επιχειρήσεις Βρετανικές, να φύγουν την Τελωνική Ένωση του 19ου αιώνα και να μπουν σε ένα κλίμα πιο απελευθερωμένο, πιο επιχειρηματικό αλλά δυστυχώ τα βλέπει διαφορετικά η ε, Πρωθυπουργό μα, αλλά μάλλον θα ιτηθεί ε, και θα ταπεινωθεί σήμερα και θα το απολαύσω και ελπίζω ότι θα βγούμε σύντομα την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνάψουμε συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου με τον υπόλοιπο κόσμο. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, το πρόγραμμα InvestEU για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που ακολουθεί θα ε, χρηματοδοτήσει πολλά προγράμματα. Εσείς μιλήσατε για 13. Θα υπάρξει ε, μεγαλύτερη ευελιξία. Ε, ολοκληρώνεται το 2021 και το δεύτερο επενδυτικό σχέδιο και θα κλείσουν και κάποια κενά επενδυτικά τα οποία έχουν παραμείνει. Έχουμε και τα 38 δις. Εμείς θέλαμε 40 αυτά στο πλαίσιο της εγγύησης αυτής. Ε, συνολικά θα κινητοποιηθούν 50 δις και πιστεύω ότι έτσι ε, θα έχουμε κάποια πρόοδο. Σίγουρα ε, η ε, εξυγίανση έχει βοηθηθεί και από την ΕΤΕΠ θα έχουμε το 75%. Σίγουρα και η Τράπεζα Επενδύσεων, η Μπέρντ συμμετέχουν, η Παγκόσμια Τράπεζα και Έχουμε και τα Central Advisory Hubs και τους εταίρους αυτών. Ε, τα 650 δις ε, στους τέσσερις τομείς ε, για το έτσι για το InvestEU είναι θετικό. Ας ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές. Παύλο Ρούμπιχ τώρα έχει το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω ε, και τον ε, Βίλ Μόρτεν που, που έδειξε πόσο μπορούμε να ε, εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα και ο κύριος Κατάινεν ε, έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Σίγουρα οι επενδύσεις πήγαιναν πίσω, ε, θέλαμε το 20% να πετύχουμε, είμαστε σε 15%, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία είναι στο 10%. Άρα βλέπουμε ότι ε, χρειάζεται ακόμη να δράσουμε. Εγώ μέχρι το 2030 θα έλεγα ότι το 30% της παραγωγής θα έπρεπε να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σημαίνει ότι θα πρέπει να προσελκύσουμε ε, την παραγωγή, η οποία έχει μετεγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια σε τρίτε χώρε, ε, να την προσελκύσουμε λοιπόν ε, με τη βιομηχανία 4.0 και με τη ιδέε μέτρων για τι δεξιότητε και όλα τα άλλα μέτρα τα οποία έχουμε προωθήσει. Και αυτό το SME Window είναι κάτι που πρέπει να το αξιοποιήσουμε και για τον επιμερισμό των κινδύνων. Χρειάζεται ανάληψη κινδύνων και από τι μικρομεσαίες και τις μεσές επιχειρήσεις και φυσικά οι μεγάλες επιχειρήσεις. Το 5% και πάνω του ΑΕΠ είναι από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάρα πολλές θέσεις εργασίας παράγονται από τις, και προσφέρονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουμε αυτό το 75% των, ε, που θα τροφοδοτείται από την ΕΤΕΠ και το 25% από τις Εθνικές Τράπεζες είναι κάτι καλό και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα πολύ καλύτερο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπερές έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό από τους Αστές Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βελτίωσε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαιρόμαστε ιδιαίτερω γι' αυτό. Γιατί είναι σημαντική αυτή η πρόταση για να δώσουμε μια νέα όθηση στι ε, επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πραγματικά υπήρχε μεγάλο κενό και τι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Είναι σημαντικό για του πολίτε, για τι επιχειρήσει και για τι περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι για την προσπάθεια πλούστευση των τρόπων χορηγιστών επενδύσεων και να και να εξασφαλιστεί συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα και με την πολιτική συνοχή. Αυτό είναι σημαντική πρόοδο, κατά τη γνώμη μου, στην τελευταία πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά του ε, στόχου των επενδύσεων που έγιναν δεκτοί, ε, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό τη στρατηγική θα πρέπει να είναι η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συνδυάζει στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, τη Συμφωνία των Παρισίων, χωρί να μελεί τι κοινωνικέ επενδύσει και της ε, τον πολιτιστικό κλάδο και τον κλάδο της δημιουργίας. Επίσης, ε, ο συνδυασμός ε, της ΤΕΠ με τις Εθνικές και Περιφερειακές Τράπεζες Προώθησης θα βελτιώσει την κατάσταση και θα επενδύσει εκεί που χρειάζονται με χρήσιμο τρόπο ώστε να έχουμε πραγματικά καλύτερη ανάπτυξη, βιώσιμη, που θα δημιουργεί και θέσεις απασχόλησης. Από το ECR το λόγο Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, είναι το πρώτο θέμα που έχω αναλάβει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ μέρους ε, του κόμματός μου του NVA στην ομάδα των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Δεν ρωτώ με είναι χρήσιμη αυτή η πρόταση παρόλο που νομίζω ότι η προτινόμενη μεταρρύθμιση είναι αρκετά λογική. Ο συνδυασμό όλων των επενδυτικών προγραμμάτων ε, σε ένα ενίο πρόγραμμα είναι μια πολύ καλή ιδέα. Αυτή η απλοποίηση ε, είναι σωστή. Η αρχική πρόταση είχε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά το ρόλο της ε, ΕΚΤ και τη διακυβέρνηση. Αλλά σωστό είναι που δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου των εθνικών τραπεζών επενδύσεων. Ε, έτσι μπορούν να λάβουν πλήρως τα κρατημένη την ευθύνη για τον τρόπο εφαρμογή των επενδύσεων. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές για το έργο τους και το όραμά τους. Ο κύριος Σολέ έχει το λόγο, παρακαλώ, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρεις πτυχές ε, του προγράμματος InvestEU. Καταρχήν υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη κινητοποίησης ε, ε, ιδιωτικών και κρατικών κονδύλων για τι επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, οι επενδύσει θα πρέπει να έχουν μια λογική, θα πρέπει να εξυπηρετούν ένα σωστό στόχο και να εξυπηρετούν κοινού σκοπού. Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να είναι χρήσιμο εργαλείο για τη μεταμόρφωση, το μετασχηματισμό των οικονομιών μα ε, σε οικονομίε ουδέτερε ω προ τον άνθρακα και χωρί αποκλεισμού. Θα πρέπει να λάβει υπόψη την ενεργειακή μετάβαση και κλιματικού και κοινωνικού όρου και προβληματισμού. Επίση, θα πρέπει να μην υπονομεύσουμε τη Συμφωνία των Παρισίων και να υλοποιήσουμε και του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό θέλουμε πιο φιλόδοξου στόχου ε, τι δαπάνε για το περιβάλλον σε ό,τι αφορά τι στρατηγικέ επενδύσει. Θα πρέπει να αποκλειστούν επίση προγράμματα που θα μπορούσαν να είναι επιζήμια από περιβαλλοντική άποψη. Δεύτερον, είμαστε κατά τη χρηματοδότηση των αμυντικών προγραμμάτων από το InvestEU. Η στρατιωτικοποίηση του κοινοτικού προπολογισμού μέσω τη στήριξη τη έρευνα ή μέσω επενδύσεων δεν είναι ο κατάλληλο τρόπο για να επιλύσουμε τι προκλήσει ασφάλεια που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κονδύλια του InvestEU θα πρέπει να επενδύονται σε άλλου τομεί γιατί εκεί χρειάζονται πολύ περισσότερες επενδύσεις, όπως στην κοινωνική οικονομία, για παράδειγμα. Τρίτον και τελευταίο. Θέλουμε ισχυρότερη συμμετοχή ε, όχι μόνο των εθνικών, αλλά και των περιφερειακών τραπεζών πρόθεσης. Ε, έτσι θα γίνει μια καλύτερη κατανομή των σχεδίων ανάλογα με τι τοπικές ανάγκε και τι κοινωνικέ ανάγκε των τοπικών παραγόντων και φορέων. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, από το σχέδιο Juncker πήγαμε στο FC, στο FC1, FC2 και τώρα έχουμε ένα νέο όνομα, το Invest EU. Αλλάζει το όνομα, αλλά η βασική η αρχή είναι η ίδια. Η επένδυση καλύπτει περισσότερο τις ιδιωτικές επενδύσεις παρά τις δημόσιες. Εγώ δεν πιστεύω ότι η επένδυση τελικά θα καταλήξει στο δημόσιο τομέα. Εγώ δεν βλέπω βελτίωση ε, των δημοσίων μεταφορών για τη βελτίωση τη ζωή των ανθρώπων στην Ήπεθρο. Οι ιδιωτικοί επενδυτέ δεν θα καλύψουν τι δημόσιε υπηρεσίε. Στον τελευταίο κανονισμό, στους τελευταίους είχαμε διατάξει για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, συνεταιρισμών κλπ. Δεν είδα όμω κάποια στοιχεία να αναφέρονται εδώ και όποτε ζητώ στοιχεία για τα ζητήματα αυτά δεν παίρνω απαντήσει. Είμαι κάθετα κατά ε, χρημάτων που χρησιμοποιούνται για αμυντικούς σκοπούς και όλα εξαρτώνται από το πώς θα πραγματοποιήσουμε τις επενδύσεις. Θα πρέπει να γίνονται στο δημόσιο τομέα οι επενδύσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Ροζάτη έχει το λόγο για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σήμερα συζητούμε το πρόγραμμα InvestEU. Θα ήθελα όμως ε, να αναφερθώ για λίγο στο πρόδρομο του InvestEU στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Στρατηγικών Επενδύσεων που στέθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και η Ευρωζώνη κυρίως ε, έχει για 26 τρίμηνα συνεχή πρόοδο που είναι πολύ σημαντικό ε, επίτευγμα. Επίσης, το σχέδιο το επενδυτικό του Γιούγκερ συνέβαλε στην ανάπτυξη ε, και της δικής μου πατρίδας και της δικής μου γενέτειρας ε, χρηματοδοτώντας ε, εξυγχρονισμό χημικής βιομηχανίας και την βελτίωση της εσωτερικής ναυσιπλοείας στον ποταμό Όντρε. Επίσης, χάρη στο συνδυασμό και στη συγκέντρωση πολλών προγραμμάτων στο InvestEU, και με την δυνατότητα παροχής εγγυήσεων έχουμε ένα πολύ πιο ευέλικτο όργανο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό διάφορους όρους ανάλογα με τις ανάγκες των προγραμμάτων. Επίσης, το Ταμείο Εγγυήσεων που στηρίζει το πρόγραμμα InvestEU θα ήθελα να διευρυνθεί όπως προτείνουν οι συνεισηγητές στο 40,8 δισεκατομμύρια. Πιστεύω ότι θα αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια και χρειάζονται. Επίσης, θα ήθελα το Ταμείο σε μεγαλύτερο βαθμό να λαμβάνει υπόψη τις αναπτυσσόμενες οικονομίες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοφόντα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ανοίγει το δρόμο σε περισσότερες ειδικέ επενδύσεις για την Ευρώπη, κάτι που χρειάζεται, αλλά ε, πώς θέλουμε να δαπανίσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων ε, σε σχέση με το ε, πρόγραμμα InvestEU Business as usual. Θα εξακολουθήσουμε να επενδύουμε απερχαιωμένες προσεγγίσεις και πρακτικές του παρελθόντος ή να επενδύσουμε σε εργαλεία του μέλλοντος, στην Ευρώπη του αύριο, όπου η ανάπτυξη δεν θα επιβαρύνει τη βιωσιμότητα και το κλίμα. Αύριο θα ψηφίσουμε και είναι ένα, θέμα πρέπει να, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το θέσουμε όλοι στους εαυτού μας. Έχουμε τη δυνατότητα με αυτό το πρόγραμμα να δείξουμε την κατεύθυνση στην οποία θέλει να στραφεί η Ευρώπη ως πολιτική. Θα Πρέπει να βάλουμε πρώτα την Ευρώπη και το κλίμα. Έχουμε φιλόδοξες προτάσει από συναδέλφου υπέρ τη βιωσιμότητα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδίως ε, τους συντηρητικούς συναδέλφους ε, ε, και να τους ζητήσω να ψηφίσουν υπέρ ενός προγράμματος που θα βάζει το κλίμα και το μέλλον στην, ως προτεραιότητα στην κορυφή. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό κυρία Τιλιμέτς. Ε, ε, Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, για μένα το κεντρικό σημείο του προγράμματος InvestEU είναι ε, να συνεχίσουμε να γυρίζουμε την πλάτη σε πολιτικές λιτότητας, αλλά να επενδύσουμε σε καινοτόμα βιώσιμα έργα. Όμω, όμως, αν δεν υπάρχει υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα σχέδια δεν θα υποστηριχθούν. 38 δις, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι γιατί ποσό μιλάμε, για σχέδια τα οποία ε, θα προωθήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραδείγματο χάρη που δραστηριοποιεί στον τομέα της ε, παροχής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία, αεολικά, πάρκα στην βόρεια ε, θάλασσα, ενεργή, θερμική, εξοπλισμός για την θερμομόνωση στο πλαίσιο ενεργής απόδοσης των κτηρίων κτλ. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι υπάρχει και δαμόκλειο σπάθη, προσπάθεια της εξοπλιστικής βιομηχανίας να σφετεριστεί του πόρους αυτού. Πρέπει στι ειρήνε τη Βιομηχανία ε, τη εξοπλιστική να κλείσουμε τα αυτιά μας, αγαπητοί συνάδελφοι, για να εξασφαλίσουμε το μέλλον του πλανήτη Μα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Φανίστελ Ρόι τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Thank you, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Του συζητητέ, κύριε Επίτροπε Καϊτάνεν, συνάδελφοι. Ήδη έχουμε κάνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια του σχεδίου Juncker. Με τα χαράς βλέπω ότι κάποιες από αυτές τις αλλαγές έχουν ληφθεί υπόψη. Κάποιε επιθυμίε ελήφθησαν υπόψη. Καλύτερη σχέση Φερρυπίν με την περιφερειακή πολιτική, καλύτερο συσχετισμό με τα θετικά ταμεία και με τον ορίζοντα Ευρώπη, το Horizon Europe. Μπορούμε να έχουμε περισσότερη ορατότητα και αποτελέσματα αν συνδυάσουμε αυτού του πόρου με το νέο πλαίσιο, το νέο ταμείο Invest EU για να δώσουμε μεγαλύτερη ορατότητα της Ευρώπης προς πολίτες. Δεύτερον, να μεταφέρουμε πόρους από τα μία. ταμεία. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του κανονισμού. Σημαντικότατο αυτό είναι ελεύθερη αυτή η μεταφορά και μπορεί να γίνει βάση ε, προτεραιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Τρίτον, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει, οι συμβουλές βοηθούν είναι απόλυτα αναγκαία στοιχεία σε όλη την Ευρώπη. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να συνεργαστεί με άλλου εταίρου σε εταιρικέ σχέσει. Τελευταίο σχόλιο. Η γεωγραφική ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα από ό,τι πριν. Δεν είναι καλό ένα μέρος της Ευρώπης να παίρνει ε, να χάνει πολλού νέου που πηγαίνουν, μεταναστεύουν αλλού, άλλο μέρο τη Ευρώπη να βρουν δουλειά. Στόχο μα στην Ευρώπη είναι να έχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη. Και νομίζω ότι ελήφθη υπόψη και καλύπτεται καλύτερα. Σαν συντονιστή τη Ρέτζη, υποστηρίζω την πρωτοβουλία σα. Είναι κάτι καλό για μια ε, αναπτυσσόμενη πράσινη Ευρώπη με θέσει απασχόληση. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία προσέγγιση προσέγγιση του Προέδρου. Ο κύριος ε, Μάτο Μαριά, Βιέγκας, Μάλετη, Τσουισνέσκα, αυτοί είναι οι συνάδελφοι. Ο κύριος Γκάμπριελ Μάτο είναι ο πρώτος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω το πρόγραμμα InvestEU που σε τελική ανάλυση αυτό που ζητάει είναι η χρηματοδότηση για επενδυτικά προγράμματα στην Ευρώπη να είναι απλούστερη, πιο αποτελεσματική και πιο ευέλικτη, πιο ελαστική. Μιλάμε για επενδύσει 650 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ χαρμόσυνη ειδήση για όλου και νέα ευκαιρία για να τονώσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, την έρευνα και την καινοτομία. Βέβαια, τέτοιε ευκαιρίε θα πρέπει να ωφελήσουν και τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ, ε, ε ξεπερνώντα τα εμπόδια που ε, αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές για την πρόσβαση στις επενδύσεις. Οι, τα Κανάρια νησιά θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να λεφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Κανάριων νήσων. Η αλληλεγγύη είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην περίπτωση αυτή οποιαδήποτε εξαίρεση υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών έχει ε, την υποστήριξη, τη νομική βάση του άρθρου 349 της Συνθήκης. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. το investeu μπορεί να αποδειχθεί ένα θετικό πρόγραμμα υπό τον όρο ότι θα τεθούν ορισμένες προϋποθέσεις. πρώτον πρέπει να στηριχτούν οι απόκεντρες περιοχές και ιδίως τα νησιά του αιγαίου. δεύτερον να στηριχτούν οι περιφέρειες και όχι το κέντρο του σκληρού πυρήνα της ευρωζώνης. τρίτον να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. αυτές είναι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μια διαφορετική κατεύθυνση οι τομείς στους οποίους πρέπει να ασχοληθούμε οπωσδήποτε ο πολιτισμό, η προστασία του περιβάλλοντος η ενίσχυση της απασχόλησης. δεν πρέπει να αξιοποιηθούν τα χρήματα προκειμένου να έχουμε περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής ένωσης και κυρίως δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα που δίνει το σχέδιο juncker διότι στην ελλάδα τα χρήματα τα οποία ήρθαν επί του πρακτέου χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου η fraport να αγοράσει τα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια και δεύτερον να χρηματοδοτηθεί η κοσμοτέ η οποία είναι μια επιχείρηση γερμανική. ας έρθουν τα χρήματα στην ελλάδα για να στηριχθούν και ελληνικές επιχειρήσεις όχι οι πολυεθνικές. ας αποφύγουμε λοιπόν το κακό παράδειγμα που είχαμε στο σχέδιο juncker. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βιέγκας έχει το λόγο από την ΚΟΕ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα αυτό έχει δύο προβλήματα. Πρώτον, είναι ένα ακόμη όργανο ε, υποστήριξης του ιδιωτικού κλάδου. Υπάρχει πείνα, υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, υπάρχει φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και Αμέσω για να ενισχύσουμε τι επενδύσει, θέλουμε να στηρίξουμε τι επιχειρήσει. τον ιδιωτικό κλάδο. Αυτό δεν ανταποκρίνεται όμω στι πραγματικέ ανάγκε Ευρωπαϊκή Ένωση, στι πραγματικέ ανάγκε των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα ανταποκρίνεται στι ανάγκε του πληθυσμού και θα δίνει ε, νέα δυναμική στην οικονομία, θα τονώνει την οικονομία. Επίση, τα χρήματα που έδωσε η ΕΚΤ τα πλαίσια τη ποσοτική χαλάρωσης θα μπορούσαν να δοθούν για την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου, για να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη και να καταπολεμηθούν οι ανισότητες και οι συμμετρίες. Δεν ήταν όμως αυτό ο προσανατολισμό. Έχουμε ένα επιπλέον χρηματοδοτικό ανταγωνιστικό